στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι η παρεμβάσει διαρκείας ενός λεπτού βάσει του άρθρου 150 του κανονισμού. Έχουν ζητήσει το λόγο κάποιοι συνάδελφοι και θα σας παρακαλέσω να παίρνει το λόγο ένας μετά τον άλλον. Πρώτος ο κύριος Άνταμ Κόσακ. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Άνταμ Κόσα, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει και το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό έχει να κάνει και ε, με ε, ανθρώπους και άτομα με αναπηρίες. Θέλω να σας πω ότι βάσει του χάρτη αυτού δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις έμεσες ή άμεσες εις βάρος ε, προσώπων με αναπηρία. Είτε πρόκειται για παιδιά, είτε πρόκειται για ενήλικες και δεν επιτρέπεται πλέον καμία ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί, να ασφαλίσει κάποιον ενδιαφερόμενο επειδή έχει μια αναπηρία. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, βάσει και των δικών μας αξιών των χριστιανοδημοκρατών θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι και τα άτομα με αναπηρίες να έχουν τη θέση τους στην κοινωνία και να τους αντιμετωπίζουν όλοι με αξιοπρέπεια και με εκτίμηση και με σεβασμό. Αυτά ήθελα να σας πω και να σας παρακαλέσω να Υποστηρίξτε τη διακομματική ομάδα για άτομα με αναπηρία στην ίδρυσή της. Ε, Ευχαριστώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ένας στους 7 πολίτες είναι μέλος μειονότητας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα των μειονοτήτων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όλοι γνωρίζουν ότι η δημοκρατία κρίνεται και αξιολογείται κάθε φορά από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στις μειονότητές της. Και η συνθήκη της Λισαβόνας ε, ορίζει ε, το σεβασμό των μειονοτήτων και ο χάρτης των μελιωδών δικαιωμάτων απαγορεύει διακρίσεις και ανητικές μεταχειρήσεις στις βάρος μειονοτήτων. Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα και μιλώ για τη Λιθουανία συγκεκριμένα. Τα τελευταία 20 χρόνια πολίτες Λιθουανοί υφίστανται διακρίσεις σε διάφορα επίπεδα της ζωής στην κοινωνία και ε, μιλώ για την πολωνική μειονότητα. Ένα λεπτό, ο κύριος Γιάρος Άφολε. Αγαπητέ Πρόεδρε, στις 14 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την στρατηγική της ε, για την ε, διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Α, σε σχέση με την παγκόσμια οικονομική κρίση έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και για αυτές τις χώρες. Εις ό,τι αφορά την, Επιτροπή, την Μικτή Επιτροπή για την Τουρκία θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την πρόοδο που θα πρέπει να επιτύχει η χώρα ε, στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, και στην πολιτική καλής γειτονίας. Θα πρέπει η Τουρκία να αναλάβει περισσότερες δεσμεύσεις για να σεβαστεί τα κριτήρια. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση στις τουρκικές αρχές για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, για το ξεχρονισμό της χώρας και για την ενσωμάτωση του κεκτημένου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Μαρτυραβέλα για ένα λεπτό. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, κάθε περάσαμε το δισεκατομμύρια άτομα που υποφέρουν από υποσυτισμό. Αυτό αναφέρθηκε στη σύνοδο του Πίτσμπεργκ στον G20. 20 δισεκατομμύρια δολάρια αναγγέλθηκαν ως βοήθεια στην γεωργία και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είχε γίνει και στη σύνοδο των G8 στο Λάκουιλα, αλλά στις 16 Νοεμβρίου στα πλαίσια της ΦΑΟ η σύνοδος έδειξε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Ε, δεν κατέληξε στην επικύρωση των μέτρων που περιμέναμε κανένας, καμιά δέσμευση με ποσά δεν αναφέρεται στα 40 άρθρα, ούτε καν τα 44 δισεκατομμύρια για την υποστήριξη της γεωργίας των πτωχοτέρων χωρών που έκρινε απαραίτητα η ΦΑΟ. Απλώς χαιρετίστηκε η υπόσχεση των μελών που ήταν στην Άκουιλα για αυτό το σχέδιο. Πρόκειται λοιπόν για μια διπλή γλώσσα, για μια διγλωσία. Αμφιβάλλουμε λοιπόν για το μέτρο αυτό και όπως έλεγε ο Πιέρ Ντάκο λέω ότι χρειάζεται ατελείωτη υπομονή για να περιμένει κανείς αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντώνιο Μασίπιλντάγκο. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Αστουρίας, που είναι η περιοχή μου, αλλά και πολλές άλλες οργανώσεις ε, δακτυλοδεικνύουν την περιοχή ε, επειδή επισκέφθηκαν στο Τιντούφ τι ε, οικογένειέ του, φυλακίστηκαν άνθρωποι, πολιτικοί κρατούμενοι, βασανιστήρια, καταπάτηση του διεθνού δικαίου. Μία ηρωίδα που προσήφιε το βραβείο Ζαχαρόφ, η αμυντή του Χάινερ, ε, απελάστηκε, α, ναι, απελάστηκε από την χώρα. η κυρία Μάλστρομ και όλα τα όργανα της Ένωσης θα πρέπει να αναλάβουν δράση για τον πληθυσμό της υποσαχάριας ε, περιοχής. Ε, δεν είναι μόνο το τείχος του Βερολίνου, δεν ήταν μόνο το τείχος του Βερολίνου, υπάρχει και άλλο ένα τείχος στην περιοχή αυτή που θα πρέπει να γκρεμίσουμε. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρλ Χάγκλαντ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία βδομάδα... Ακούσαμε πολλά για την Βαλτική και θα ήθελα να πω κάτι για την Βαλτική θάλασσα. Την τελευταία εβδομάδα, την Τετάρτη, είχαμε μια συνδιαλλαγή ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει τα 20 εκατομμύρια για την στρατηγική της Βαλτικής θάλασσας που το Κοινοβούλιο πρόσθεσε στην πρώτη ανάγνωση και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια νομική βάση για την στρατηγική της Βαλτικής θάλασσας και θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό στην Επιτροπή ούτως ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια. Και βεβαίως η κατάσταση είναι κατεπίγουσα. Και ελπίζω ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι κατεπηγόντως θα πρέπει να έχουμε ε, αμέσως μέτρα από τον Κομισιό και από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, ο η κυρία Φλότρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήμουν στην Τινησία ε, για την δίκη του Ταφίκ Μπενμπρίκ, ποιητή και ανθρώπου των γραμμάτων που κατηγορήθηκε με σκοτεινούς και δόλιους τρόπους Κανείς όμως δεν απατάται από τις εκλογές στην Τινησία, από τότε που έγιναν οι εκλογές στην Τινησία, ε, ξεκίνησαν κατακλυσμίες αρνητικές ε, ε δράσεις και φαινόμενα. Ο κύριος Μπεναλή ε, κατάλαβε ε, πόσο δεν χαίρει καμία εκτίμηση από την κοινή γνώμη, αλλά όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της γενικής αδιαφορίας των πρεσβειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δυστυχώς δεν έχει αρμοδιότητες ε, και δεν έλαβε και θεώρηση, τα μέλη της δεν έλαβαν θεώρηση για να παραστούν σε αυτή τη δίκη. Τι περιμένουμε λοιπόν στις πρεσβείες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλέσουμε με το πιο έντονο τρόπο στο όνομα των συμφωνιών που έχουμε με τη χώρα. Τι περιμένουμε, λέω, για να καλέσουμε τον κύριο Μπεναλή να λογοδοτήσει για τις δράσεις του που είναι εντελώς αντίθετες με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ευχαριστώ. Βάλτε το Μασεύσκι. Ε, ε, Ο κύριος Ζωάου Φερέιρα. Η εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε στις 4 του μηνός μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ για τα γεωργικά προϊόντα και τα λευτικά προϊόντα είναι εντελώς απαράδεκτη για διάφορους λόγους, τους οποίους εδώ καταγγέλουμε. Πρόκειται για νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιτείνουν την υπάρχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση, ιδιαίτερα στη Γεωργία και την Αλία. Αυτό όμως είναι ιδιαίτερα πιο σοβαρό όταν αυτές οι πολιτικές προωθούνται μέσω, μιας, συμφωνίας με μια χώρα που παραβαίνει το διεθνές δίκαιο και τα πιο βασικά δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού και που δεν δέχεται τις ε, δεσμεύσει που έχουν αναλυθεί δυνάμει του φίλου πορεία για την ειρήνη, του οδικού χάρτη του λογομένου. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτίζει τύχη, συνεχίζει να διώκει του Παλαιστίνιου πολίτε, συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνέ κράτο δικαίου. Καταδικάζουμε την υπογραφή αυτή τη συμφωνία ε, που θα ε, αποτελέσει μία ακόμα ντροπή στη σχέση μας με το Ισραήλ, το οποίο επιτέλους πρέπει να επαναφέρουμε στην τάξη. Εκφράζουμε εδώ την αλληλική μας με το Παλαιστινιακό λαό και υποστηρίζουμε την προσπάθειά τους για ένα ανεξάρτητο, ελεύθερο και κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζέραρντ Μπάτεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ε, Ρώσος ε, εξόριστος πρόσφατα δημοσίευσε τη σχέση του, του εργατικού κόμματος α, ε, της Μεγάλης Βρετανίας με τη Σοβιετική Ένωση. Ε, απόρριτα έγγραφα λέγουν ότι το 80 ο Νίλ Κίνοκ ηγέτης της αντιπολίτευσης τότε προσέγγισε τον κύριο Γκόρμπατσοφ, έστειλε κάτι απεσταλμένους για να δει τι θα γινόταν εάν σταματούσαν τις πυρηνικές δοκιμές. Αν είναι σωστό αυτό και ισχύει η έκθεση, σημαίνει ότι ο Ρόδος Κίνοκ προσέγγισε έναν ε, ε, από τους εχθρούς της Βρετανίας για να εγκριθεί η ε, πολιτική του ως προς τα πυρηνικά και αν εκλεγόταν στην κυβέρνηση θα ήταν και η βρετανική πολιτική. Αυτό είναι σχάτη προδοσία αν ισχύει. Και θα πρέπει σε ύψιστο επίπεδο να το εξετάσουν οι αρμόδιες αγγλικές αρχές και να έρθει να απολογηθεί ο κύριος Κίνοκ για αυτά τα στοιχεία τα σοβιετικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σας θυμίσω ότι όσοι ζητούν τώρα το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχω ένα κατάλογο με 79 βουλευτές και μέχρι 30, το πολύ 35 μπορούν να πάρουν το λόγο. Υπάρχει ήδη κατάλογος, μην ζητάτε καινούργοι τώρα το λόγο. Ε, λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα έπρεπε να το είχατε ζητήσει εκ των προτέρων. Δεν μπορώ να πάρω καινούργια ονόματα τώρα. Ο κύριος Τσάμπα Σόγκορ. Ευχαριστώ. Είναι λυπηρό ότι η πολιτική των μειονοτήτων και των γλωσσών που μιλούν οι μειονότητες ε, δεν θεωρείται σημαντική στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο ε, γιατί ε, επεμβαίνει και κάνει ε, διαβήματα και στη Σλοβακία. Υπάρχουν προβλήματα στη Σλοβακία και το θέμα της γλώσσας είναι το λιγότερο. Επίσης, στη Τσεχική Δημοκρατία δεν χρειαζόταν η συνθήκη της Λισαβόνας για να δούμε τι σημαίνουν τα διατάγματα μπενές. Πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει με τη συλλογική ευθύνη και όχι με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά και αντίθετα προς το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζουμε το μέλλον της Ευρώπης ε, να μην καθορίζεται από τη συλλογική τιμωρία και τη συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά από τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν ατομικά και την αυτονομία. Κυρία Ζαμπόρσκα. E, Ευχαριστώ. Έχουμε ε, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού ε, που είναι μια σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και φέτος τον Νοέμβριο έχουμε μια επέτειο ε, και μας ενδιαφέρουν πολύ τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα της οικογένειας όσο βλέπουμε ε, γύρανση του πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με θέματα οικογενειών, με θέματα παιδιών, με θέματα ε, αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων γενεών. Ε, χρειάζονται επαγγελματίες της υγείας και επαγγελματίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να προστατεύουν τα παιδιά. Η σύμβαση λέει ότι το παιδί για να ε, μεγαλώσει καλά θα πρέπει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια, σε ένα σπιτικό που να βασίζεται στην ευτυχία, στην αγάπη, στην κατανόηση και στη στοργή. Εδώ ε, πρόκειται τώρα για μια πλατφόρμα που προτείνουμε βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες και καλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν τη διακομματική ομάδα, το Intergroup αυτό για τα δικαιώματα του παιδιού και είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί. Ευχαριστώ, Σάρμπο. εξ ε, της ε, κοινότητα, το θέμα κοινότητας των Ρώμα στην Ιταλία μας απασχολεί πάρα πολύ. Όλη η Ευρώπη γνωρίζει με ποιο τρόπο έχει κατηγορηθεί ολόκληρη μια κοινότητα λόγω ορισμένων ατόμων. Εκφοβίζεται αυτή η κοινότητα, υποφέρει αυτή η κοινότητα. Μερικά παραδείγματα. Ο τύπος ε, διηγήθηκε μια κατάφορη περίπτωση διάκρισης. Στην Ιταλία ένας οργανισμός τηλεφωνικός, ε, ο διευθυντής συνέστησε ε, στους εργαζόμενους να μην συνάπτουν συμβόλαια με ρουμανικής καταγωγής άτομα άτομα ε, σε ένα νοσοκομείο, ένα Ρώμα δεν έγινε δεκτός, δεν τον δεχόταν κανένα νοσοκομείο και πέθανε στο δρόμο. Αυτοί που βρίσκονται ε, συναντούν αυτά τα προβλήματα κάθε μέρα. Νομίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε να επισύρουμε την προσοχή της Ιταλικής ε, κυβέρνησης στο πρόβλημα αυτό, ούτως ώστε να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των Ρουμάνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επρόκειτο να μιλήσω για την ε, σημασία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για την Ιουαλία μετά το 2013. Πρέπει να απαντήσω στα σχόλια του κύριου Μπακενέλια ε, σχετικά με τον ε, πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του και ζητώ αυτές οι παρατηρήσεις να αποσυρθούν, να του ζητήσετε να αποσύρει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τα οποία έκανε. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον Ιμπο Βάιγκλ να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τι θα μας πει ο, η υποψήφια για το, τη θέση της, του υπάτου εκπροσώπου. Θα είναι και επίσης μια δοκιμασία και για μας επίσης η απάντηση στο θέμα της επίδρασης που μπορεί ε, να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής και αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν ενεργό ρόλο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πάρα πολύ επιτυχία. Ο συνάδελφος που μίλησε πριν από μένα αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ο φαύλος κύκλος στην Παλαιστίνη συνεχίζεται αυτές τις μέρες. Η Παλαιστίνη επιτίθεται στο Ισραήλ, το Ισραήλ απαντά δυσανάλογα, είχαμε πολλές απώλειες και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε ούτε καν για ένα λεπτό να ξεχνάμε ότι συνέχεια επισύρει πάνω του την προσοχή το Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Ντέιβις. Κύριε Πρόεδρε, οι στρατιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλα κράτη μάχονται και πεθαίνουν στο Αφγανιστάν. Μας είπανε ότι είναι για να είναι ασφαλής η χώρα μας, για να προστατευθούμε από την Αλκάιντα, για να μην υπάρχουν πια τα ναρκωτικά, για να προστατεύσουμε το Πακιστάν, τα δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών. Αλλά δεν υπάρχουν πια αυτά τα επιχειρήματα, δεν υπάρχει σαφή στρατηγική και δεν ξέρω τι επιτυγχάνει ο θάνατος των στρατιωτών μας. Αντίθετα, αυξάνονται οι κίνδυνοι και μας προδίδουν οι εξτρεμιστές, οι Ισλαμιστές που υποστηρίζουν τους, τους πολέμαρχους και τους εμπόρους ναρκωτικών. Εκεί που ε, όλους έχουν πεπιθήσεις αντιδυτικές, Ισλαμικές. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική. Πρέπει να συνομιλήσουμε με τους Ταλιμπάν, να προωθήσουμε την συμφιλίωση και να διευρύνουμε την σύνθεση της παρούσας κυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποσύρουμε τους στρατιώτες μας από τη γη του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Η Ιζαμπέλ Γκυρόν έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε μια συμφωνία ανάμεσα ε, στον Βελγικό κράτος και Ζεντεφ Σουέζ ε, συνάφθηκε το Οκτώβριο 2001 και συνεχίζει το μονοπόλιο μέχρι το 2015. Αυτό είναι αντίθετο προς τις πολιτικές απελευθέρωσης και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει το μονοπόλιο στον πυρηνικό τομέα και αυτό θα καταστήσει δυσκολότερα τα σχέδια ανανεωσίμων πηγών ενέργειας και των σχετικών θέσεων εργασίας. Όταν ξέρουμε ότι ο ρυθμιστής, ο ανεξάρτητος ε, θα αφήσει την παρακολούθηση σε μια επιτροπή παρακολούθηση όπου θα εδρεύει και η ZDF Σουέζ, ε, Διαρωτώ με τι θα γίνει και ελπίζω να έχει η Κομισιόν μια αντίδραση και να μπορέσει να αντιμετωπίσει προβλήματα όπου ε, κάποιος είναι ε, ταυτόχρονα ο παρακολουθών και ο παρακολουθούμενος. Ελπίζω η ε, Επιτροπή να αντιδράσει κυρίως την παραμονή της Κοπενχάγης όπου τα θέματα αυτά είναι σημαντικά των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω η Κομισιό να αντιδράσει ούτω ώστε η Pax Electrica να μην επιβεβαιώσει το μονοπόλιο ανάμεσα στο κράτος και στη GDF Suez. Ευχαριστώ. Στην Ιρλανδία τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον βαρεθεί να πληρώνουν ε, τις ζημινιές και τα σπασμένα της κρίσης του καπιταλισμού. Θα πρέπει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ε, μήνυμα αλληλεγγύης προς τους απεργούς εργαζόμενους Ιρλανδούς αύριο καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν την απεργία, να ρίξουν την κυβέρνηση και να προκαλέσουν γενικές βουλευτικές εκλογές να αποφασίσει ο λαός. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα, οι περικοπές είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι απολύσεις μαζικές, η κοινική συμμαχία μεταξύ ε, της σοσιαλδημοκρατίας και των φιλελευθέρων στο Κοινοβούλιο έδειξε ε, το τελευταίο της πρόσωπο. Διόρισαν ε, ύπατη εκπρόσωπο για εξωτερικά θέματα μια κυρία που ποτέ δεν εξελέγει. Οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να δώσουν μάχη να εμποδίσουν την φιλελεύθερη πλειοψηφία σε αυτό εδώ το σώμα να κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Ανδρέας Μέλτσερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ένα στου 7 Ευρωπαίους ανήκει σε εθνική μειονότητα, κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο, η προστασία των αυτοχθόνων μειονοτήτων ε, στην Ευρώπη οχριά. Θα πρέπει οι Βρυξέλλες να φέρουν ενώπιον των ευθυνών τους τα κράτη-μέλη. Νύπτη τα σχήρα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν αναμειγνύομαι μέσα εσωτερικά θέματα των κρατών μελών. Στην Ευρώπη δεν έχουμε ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων διεθνούς δικαίου. Ανάλογα με τη χώρα, με πολύ διαφορετικό τρόπο εφαρμόζονται αυτά. Η Γαλλία, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει εθνικές μειονότητες και στη Σλοβενία παραμένει ε, ε, μια διάταξη που στρέφεται κατά του διεθνούς δικαίου. Και στην Αυστρία υπάρχουν προβλήματα. Αυτό τι δείχνει. Υπάρχει ανάγκη ενός ευρωπαϊκού δικαίου μειονοτήτων η Ευρώπη ε, έχει αναπτυχθεί με εθνική ποικιλομορφία και αν θέλει να τη διατηρήσει χρειάζεται οπωσδήποτε ένα δεσμευτικό δίκαιο για αυτόχθονες μειονότητες. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδείξει ε, ότι την ενδιαφέρει αυτό το θέμα ουσιαστικά και δεν είναι ε, ωραία λόγια και κενά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Ο κύριος Σικέρσκι τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στις 9 Νοεμβρίου στο Βερολίνο εορτάστηκε η 20η επέτειος της πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Αυτοί οι εορτασμοί έδειξαν ότι ε, άνοιξε τότε ο δρόμος για τον εκδημοκρατισμό και την υπέρβαση του διχασμού όχι μόνο στη Γερμανία, σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί να ήταν η ε, ε, αφορμή ε, ή το γεγονός αυτό στο Βερολίνο, αλλά η κατάσταση συνεχίστηκε και αλλού. Το 90, α πούμε, στις πολωνικές ακτές με τη παρουσία του Βαλέσα. Για να μην πάω πιο μακριά, το 56 στην Ουγγαρία ή το 68 στην Τσεχοσλοβακία ή στο Πόσνα, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν ε, πολλοί αντιφρονούντες, ε, θαραλέοι και ενεργοί σε όλα αυτά τα κράτη που ε, αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία και μερικοί από αυτούς θυσίασαν και τη ζωή τους τότε. Τους τιμούμε, τους τιμόμαστε και όχι μόνο εκείνους και όλους τους πολιτικούς που βοήθησαν στον εκδημοκρατισμό και στη μετάβαση στη δημοκρατία. Ο Πρόεδρος, συνάδελφοι, έχω μία ανακοίνωση που θα σας αναγνώσω στα ε, αγγλικά ίσως είναι πιο εύκολο για σας. Ο κύριος David Μάρτιν έχει καθυστέρησει την πτήση του και έχουμε την έκθεσή του. Η πτήση του έχει καθυστερήσει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, αν συμφωνείτε, ε, να συζητήσουμε